Bene. Bene, iniziamo subito il voto. Mi scuso con i colleghi per qualche minuto. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η συζήτηση όπως είδατε κι εσείς σημαδεύθηκε από τη συμμετοχή πάρα πολλών συναδέλφων. Υπήρξαν άνω των 25 ομιλητών και δεν μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε τους χρόνους περισσότερο. Θα πάμε γρήγορα από εδώ και πέρα και δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση το Σενόσκι Eh, eh. ah, θα υπάρξει έλεγχο τη ηλεκτρονική ψηφοφορία για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει. Ξεκίνησε η συνεδρίαση, η ψηφοφορία, συγγνώμη, ψηφίστε παρακαλώ. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία, Πέρα της ψηφοφορίας. 45 παρόντες. Η Πιλάρα, έχει δει το λόγο, όχι λέει η Πιλάρ. Λοιπόν, εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 108. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Λοιπόν, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 22, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 14 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 12 της ΙΝΚΟ. Τέλος της ψηφοφορίας. 15 υπέρ 11 κατά δεκτή. Τροπολογία 112, 120 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά θα το ελέγξουμε παρόλα αυτά. Για την 29 πολιτισμός. 35 υπέρ δεκτή, 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 123 για συγγνώμη, 123 επαναλαμβάνει πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 125 Αφέλετε θέλετε έλεγχο για την 128. Ψηφίζετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή η τροπολογία. Παρακαλώ δείξτε μου το σημείωμα. 125 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 129 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 131 παρακαλώ απορρίπτεται με μικρή διαφορά 21-23. Λοιπόν, 132 υπέρ. Με προφορική τροπολογία η 132 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές η 14 της ίνκο Τη ΣΥΜΚΟ 14 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 14. Πέρα τη ψηφοφορία. 20 υπέρ 25 κατά πράγματι απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 159 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 160 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 161 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 165 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 169 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές Ας δοκιμάσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την 23. Ψηφίζουμε λοιπόν την 23 περιφερειακή. 29 υπέρ 15 κατά δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 172 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 172 πέρας της ψηφοφορίας. 21 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται. Λοιπόν, 173 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 35. Κοιτάξτε, οι συνδυασμοί είναι δύσκολοι σήμερα. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή η 35. 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 και 177 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές. 179 ψηφίσαμε την 22 με την 177 από κοινού και περνάμε τώρα στην 179. Εντάξει. Λοιπόν, 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μαζί την 23, την 180 και την 181 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές Φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές φαίνεται ότι απορρίπτεται θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 26 Ψηφίζουμε την 26 πέρα της ψηφοφορίας. Πάλι έλεγχος εξ αρχής για την 26. Ψηφίζουμε την 26. Τέλος. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 185 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 186 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 187 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 194 τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 206 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 20. Πέρα της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 24 κατά, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 218 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 218. 18. Respinto. 43. Λοιπόν, απορρίφθηκε. Δεν είχατε σηκώσει τα χέρια σας, εδώ αριστερά δεν σας βλέπω έτσι και αλλιώς. 29 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 225 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 226 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 31 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 και 17 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 244 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ομαδών τώρα από τη 245, 46, 47. Και είναι υπέρ. Α, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος και 248. Λοιπόν, τέσσερις τοπολογίες. Όχι λένε από την αίθουσα. 245 λοιπόν, 246 και 47 από κοινού εντάξει, ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 248 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Έλεγχος για τη 248. Τέλος της ψηφοφορίας απερίφθη. 250 υπέρ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 249 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 251 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος, όχι, ε, απερίφη, εύκολα, αλλά υπάρχει έλεγχος εφόσον το επιθυμείτε. Ψηφίζουμε. πέραστη της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 30 κατά. Συμβιβαστική 33 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 2.55 Α, όχι, συγγνώμη. Έχει αποσυρθεί η 2.55. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 34. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2.57 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 35 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 262 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 263 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά Δεκτή 43, 36 και 2,65 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 269 υπέρ. Με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 21. «24 υπέρ 22 κατά γίνεται δεκτή». Συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 272 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 273 υπέρ κατά αποχές δεκτή μαζί 274 και 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.80 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε ομαδών από την 83 μέχρι την 89. Όλες μαζί. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 44 και 18 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 290 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 291 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή μαζί την 7 και τη 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 και 66 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 8. Αρχίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10 και 4 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77-78 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ και 6 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές, απορρίπτονται μάλλον, συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 82 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 88 υπέρ κατά αποχές δεκτή 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 και 90 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 και 100 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή. 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 102 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 20 και 8 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 107 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τελική ψήφος ηλεκτρονική. Votazione chiusa. Πέρα της ψηφοφορίας. 44 υπέρ 1 κατά. Ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Ποιοι είναι υπέρ. Πέρα της ψηφοφορία 44 υπέρ 1 κατά μία αποχή. Πολύ καλά. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και περνάμε τώρα στην έκθεση Κόβατς. Α, όχι, λάθος λέει η πρόεδρος. Κόβατς. Porto Κόβατς, noi qui abbiamo soltanto un voto soltanto un voto sulla legislativa, votazione aperta sul rapporto Kovac, prego. Votazione chiusa. Bene, 39 a favore. 39 υπέρ, 1 κατά μία αποχή δεκτή για την έκθεση Κόβατς. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση Χέντσου. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία στη συμβιβαστική 2 για την έκθεση έντσιου. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία έντσιου. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ λέει ο κ. Έντσιου. θα πρότεινα να διαγραφεί η αναφορά στις μη, μη συμβατικές ενεργειακές πηγές. Το είχα ήδη προτείνει. Δεν ξέρω γιατί το κείμενο δεν άλλαξε. Η τροπολογία είναι πολύ απλή. Προτείνω τη διαγραφή της λέξης non-conventional, μη συμβατική, μη συμβατικές. Αν θέλετε μπορώ να σας το διαβάσω κιόλας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 Πηγές ενέργειας, να λέει στο τέλος, όχι μη συμβατικές πηγές ενέργειας. Θέλω να διαγραφεί η λέξη non-conventional. Εφόσον συμφωνείτε, λέει πρόεδρος, πάνω στην προφορική τροπολογία NCU. Λοιπόν, ψηφίζουμε την συμβιβαστική 2. Είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 είπε. κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 17 παρακαλώ. Τέλος της, της ε, ψηφοφορίας 21 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχής δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψήφος άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική θυμίζω. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας, 43 υπέρ, 1 κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια. Περνάμε στην έκθεση Λάγκεν. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 58 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ και 68 από κοινού. 66 και 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 65, 66, 67 και 70 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 και 10 α όχι μια στιγμή διορθώνει πρόεδρος μόνο 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Κοιτάξτε, ψηφίσαμε την 10. Τώρα θα ψηφίσουμε την 11. Θα ξαναγίνει η ψηφοφορία λοιπόν για την 11. Αν πρέπει να ψηφίσουμε και την 72, διαρωτάται η πρόεδρος. Ναι, λάθος, λάθος, λάθος. Πάμε πίσω λοιπόν. Ψηφίσαμε λοιπόν την 71, την 10 και τώρα θα ψηφίσουμε την 72. Λοιπόν, 72, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές δε, απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 88 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19, 93 μαζί υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 και 97 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20, 99 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 και 100 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές 98 α, συγγνώμη 25 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 και 103 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110-111 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά δεκτή. 116 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 <coughs> υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 42 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 129 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 130 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 131 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 133 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 134 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 130, ή μάλλον 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 100, ή μάλλον 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 138 υπέρ, κατά, αποχές, δε, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 139 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 49 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 140 υπέρ, κατά, αποχές, δε, απορρίπτεται, 141 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 50 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 142 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 51, 51 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 143 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 144 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τι έγινε με την 135 λέει Πιλάρ. 135. Ok, ok, no problem. Ok, bene. Allora siamo a posto. Voto finale. Λοιπόν, φτάσαμε στην τελική ψήφο για την έκθεση Λάγκεν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 37 υπέρ 6 κατά 3 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Για τα stress test, τα τεστ κοπόσεως υπέρ. Τέλος της ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Για τη βιομηχανία προφορική ερώτηση υπέρ. Τέλος, ομόφωνα και εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας, για την ψηφοφορία. Στην αρχή είχαμε κάποια προβλήματα, είχα κάποια προβλήματα, μετά πήγα καλά. Λοιπόν, επόμενη συνάντησή μας είναι 27 Νοεμβρίου, όπου θα έχουμε και την προσανατολιστική ψήφο λεγόμενη. Λοιπόν, σε πέντε λεπτά συνεδριάζουν οι συντονιστές. Και για παρακαλώ όσοι δεν θα καθίσουν στη συνεδρία να φύγουν από την αίθουσα.